everybody. Uh, a very warm welcome to our um, special meeting of the Internal Market Committee this afternoon. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής μας. Έχω τη χαρά και το προνόμιο να είμαι σε θέση να καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την κυρία Ινέ Στάνενμπαουμ, που είναι πρόεδρος της ε, Επιτροπή, ε, Προστασία των Καταναλωτών και Ασφάλισης Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ και θα αφιερώσουμε όλη τη συνεδρίαση στι συζητήσει μας με την κυρία Τέρνμπαουμ. Θα μας κάνει την εισαγωγή τη παρουσίαση και στη συνέχεια θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις και είμαι βέβαιο ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνεδρίαση. Μπορεί να γνωρίζουν πολλά μέλη τη Επιτροπής μα ότι σχέσει μας με την Επιτροπή αυτή και την Πρόεδρο τη ξεκίνησαν από την περασμένη θητεία ε, με την Αννίν Μακάρθη, καλή ε, συνάδελφο και φίλη που τότε ήταν πρόεδρος της Επιτροπής μας. Ε, είχαμε μεταβεί και στο Μέριλαν των Ηνωμένων Πολιτειών στην έδρα της Επιτροπής το 2008 σε επίσημη επίσκεψη και η κυρία Μπαουμ στη συνέχεια έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διατηρούμε τις επαφές και τις σχέσεις μας και τις εμβαθύνουμε και με τηλεδιάσκεψη που είχαμε πριν από λίγους μήνες, η κυρία Τένμπαμ και εγώ, Και, ε, ε, στη συνέχεια λοιπόν την προσκαλέσαμε και χαίρομαι που τόσο γρήγορα δέχτηκε και ε, κατάφερε και σε ένα πρόγραμμα μιας εβδομάδας στην Ευρώπη να βρει χρόνο να έρθει και στην Επιτροπή μας. Η Ισπανική Προεδρία ενδιαφέρεται πολύ για την προστασία των καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, επίσης, με χαρά θα καλωσορίσω ε, τον κύριο Βίτο Μορέιρα που είναι πρόεδρος της ε, Αδελφής Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και ενδιαφέρεται και εκείνος πάρα πολύ ε, για τις εργασίες μας αυτές, για τα θέματα που μας απασχολούν. Συνεργαζόμαστε συχνά ε, στη διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών που είναι σημαντικό όργανο του Κοινοβουλίου και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις εργασίες των Επιτροπών μας και να εργαζόμαστε όσο γίνεται καλύτερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και εσάς σήμερα εδώ παρόντα. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσουμε κάποιες εξελίξεις από την περασμένη συνάντηση που είχαμε με τον προκάτοχό σας. Γιατί γνωρίζω ότι στο Κογκρέσο το 2008 εγκρίθηκε ένα σημαντικός νόμος για την προστασία των καταναλωτών έχουν μεσολαβήσει λοιπόν σημαντικέ εξελίξεις και ξέρουμε ότι συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ ε, αντιθήκατε με την κυρία Σεντόρη και αργότερα θα έχουμε και δείπνο με ε, τον αρμόδιο επίτροπο θέλουμε να ακούσουμε και τις σκέψεις σα για το τι συμβαίνει στην Κίνα, την παραγωγή διαφόρων καταναλωτικών αγαθών, παιχνιδιών κτλ. Και αυτό ε, θα έχει κάποιο ενδιαφέρον και όπως γνωρίζετε συνεργαζόμαστε πάρα πολύ νερά αυτό τον καιρό για θέματα τυποποίηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο και ο κύριος Μωρέ ενδιαφέρεται πάρα πολύ από την δική του επιτροπή. Έτσι λοιπόν, τα λέω αυτά προκαταρκτικά. Θα σας παρακαλέσω τώρα να λάβετε το λόγο και μετά να ακούσουμε τις ερωτήσεις των συναδέλφων μου, καθώς επίσης και από τον κύριο Μωρέιρας. Αρκούμε σε αυτά λοιπόν και σας παρακαλώ να λάβετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ τον Πρόεδρό σας για την ευγενική του εισαγωγή. Ευχαριστώ επίσης για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας απευθύνω το λόγο στο το πραγματικά εντυπωσιακό χώρο. Ο πρόεδρος Ομπάμα ανέθεσε σε ένα μικρό οργανισμό ένα τεράστιο καθήκον, την προστασία των Αμερικανών καταναλωτών από επικίνδυνα προϊόντα. Η μακρά μου σταδιοδρομία στη Νότια Καρολίνα μέχρι να φτάσω ε, επικεφαλή του οργανισμού αυτού μου επιτρέπει να συνεχίσω να υπηρετώ το πάθος αυτό για την προστασία των παιδιών από επικίνδυνα παιχνίδια και να το επεκτείνω για να ε, προστατεύσω όλους τους Αμερικανούς καταναλωτές. Εμείς στη CEPC e οθούμεθα από αυτό το πάθος για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από οποιουσδήποτε κινδύνους που έρχονται από καταναλωτικά προϊόντα. Η επιτυχία όλων μας θα μετρηθεί από τις ζωές που θα σώσουμε, και από τους τραυματισμούς που θα βοηθήσουμε να αποφευθούν. Αυτά πέραν των ΗΠΑ και πέραν της Ευρώπης ακόμη. Ο Κόφιαναν, πρώην Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων έλεγε ότι πρέπει να είναι κοινέ οι αξίες της παγκόσμιας κοινωνίας και όλοι να υποφεληθούν από την παγκοσμιοποίηση. Και λέει, είπε ακόμη ότι θα πρέπει να επιτύχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στο βραχυπρόθεσμο κέρδος από την παγκοσμιοποίηση και μια παγκοσμιοποίηση που να έχει ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Έτσι έρχομαι στις Βρυξέλλες. Πέρασα από τη Σιγκαπούρη, το Πεκίνο, το Χονγκ και το Ανόη πρέπει να βάλουμε ανθρώπινο πρόσωπο σε αυτούς που φτιάχνουν τις παγκόσμιες αγορές, που τις ρυθμίζουν και εν τέλει καταναλώνουν τα προϊόντα της. Όσο περισσότερο εξοικειωμένοι είμαστε με τις προθέσεις των άλλων, τόσο μεγαλύτερη ευθύνη έχουμε να εναρμονίσουμε τις ευθύνες αυτές και να μεγιστοποιήσουμε την ασφάλεια να είναι γνωστοί οι κανόνες που πρέπει οι βιομηχανίε μα να ακολουθούν. Εφόσον εξοικειωμένοι με οι βιομηχανίε με αυτού του κανόνες, θα παράγουν και ασφαλέστερα προϊόντα. Ο οργανισμός μας θέλει να περιλάβει ρυθμίσεις ασφάλειας και αυτό προέρχεται από τις ε, εμπειρίες μας 2006 και 2008, όπου είχαμε διαπιστώσει ότι χρειάστηκαν κατ' επανάληψη αποσύρσεις μεγάλων ποσοτήτων παιχνιδιών που αποδείχθηκε επικίνδυνα. Και επειδή περιείχαν σημαντικά, σημαντική περιοχτικότητα μολύβδου, αλλά και επειδή ήταν εύκολο να καταποθούν. Η Κίνα είχε βρεθεί τότε στο μάτι του κυκλώνα. Όσοι θυμάστε τις αποσύρσεις αυτές θα θυμάστε ότι υπήρχαν ε, σφάλματα στην παραγωγή, σφάλματα στην αλυσίδα διανομής και επίσης δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσει ασφαλεία. Μα τι άλλαξε θα με ρωτήσετε τώρα στον οργανισμό μας. Η απάντηση είναι διπλή. Αφενό περάσαμε από, την, από το νόμο του 2008, ότι μάλλον ψηφίστηκε ο νόμος του 2008, αλλά άλλαξε και η φιλοσοφία, η ρυθμιστική φιλοσοφία. Ο νέος νόμος προκάλεσε αλλαγή παραδείγματος, όπως λέγεται και επομένως θετικές αλλαγές υπέρ του καταναλωτού. Θα σας πω ποια είναι τα χαρακτηριστικότερα σημεία του νόμου που ψήφισε το Κογκρέσο για το CPSIA και κάποιους από τους νέους κανονισμούς και ρυθμίσεις που θεσπίζουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας δούμε πρώτα το νόμο για τη βελτίωση της ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων. Ο νόμος αυτός επέφερε σημαντικότητες μεταρρυθμίσεις και διπλασίασε τον προϋπολογισμών μας και επέβαλε στον οργανισμό μας ανέθεσε στον οργανισμό μας περισσότερες ευθύνες για την παρακολούθηση της ασφάλειας των καταναλωτών για διάφορα προϊόντα τα οποία απευθύνονται στα παιδιά. Απαιτεί έρευνες από τρίτους φορείς και επίσης για προϊόντα τα οποία δεν, είναι, δεν απευθύνονται στα παιδιά και απαιτεί από τον CPSC e υποχρεωτική εφαρμογή των ε, προδιαγραφών για τα παιδιά που γνωρίζετε ποια είναι. Έχουμε, χρειάστηκε λοιπόν να εφαρμόσουμε τα standards αυτά. Επίσης τα αναθεωρούμε και εάν δεν είναι επαρκή τα κάνουμε πιο αυστηρά. Απέτησε ο νόμος αυτός ακόμη να, ε, χρησιμο... να ε, επιβάλλουμε τέτοιες ρυθμίσεις και για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε παιδικούς σταθμούς, όπως ε, καρεκλάκια, κρεβατάκια κτλ. Με επιβαλλόμενες ρυθμίσεις, εμείς εξετάσαμε την αγορά και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν 24 τομείς οι οποίοι χρειάζονται υποχρεωτικές ρυθμίσεις. Και εξετάσαμε πρώτα τις ρυθμίσεις αυτές και αν δεν είναι επαρκώς αυστηρές τότε τις κάνουμε αυστηρότερες και υποχρεωτικές. Ο νόμος ζήτησε, απίτησε από, την, από τον οργανισμό μας να παρακολουθεί την εξέλιξη των προϊόντων αυτών. 30 εκατομμύρια, προϊό... 30 ε, δολάρια ε, δαπανούμε για να φτιάξουμε μια τράπεζα δεδομένων για να βελτιώσουμε τα ε, συστήματα πληροφορικής μας, ώστε να μπορούν αυτά να επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά και να επικοινωνούν και με τα άλλα Υπουργεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ε, θα έχουμε, έχουμε μάλλον από το Μάρτιο του 2010 και μια τράπεζα δεδομένων online. Επομένω, αν κάποιο καταναλωτή έχει κάποιο πρόβλημα με ένα συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να εξετάσει και στην τράπεζα δεδομένων, αλλά μπορεί και να έρθει σε επαφή και μαζί μα για να δει ποιε είναι οι εμπειρίε μα. Αυτή τη στιγμή ανέλαβα την Προεδρία τη Επιτροπή πέρσι τον Ιούνιο Πέρασαμε ολόκληρο σχεδόν το χρόνο συντάσσοντας νομοσχέδια για τη βελτίωση της ΥΠΕΣΑΕ. Υπήρξαμε πολύ δραστήριοι για να εκπαιδεύσουμε και τους ε, ενδιαφερόμενους στο τι απαιτείται. Αλλά έχουμε συνεργαστεί και με ξένες κυβερνήσεις για να διασφαλίσουμε ώστε οι κυβερνήσεις των χωρών όπου έχουν την έδρα τους η παραγωγή να γνωρίζουν τι σημαίνει η ασφάλεια για μας. Έχουμε προτείνει και έναν ορισμό για το προϊόν που απευθύνεται σε παιδιά και αυτό μπορείτε να το βρείτε και στον ιστοχώρο μας. Οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν τι είναι παιδικό προϊόν. Ο κανονισμός λοιπόν αυτός ορίζει τι είναι παιδικό προϊόν και ότι είναι σχεδιασμένο πρωταρχικά και προορίζεται πρωταρχικά για ε, παιδιά μέχρι ηλικία 12 ετών. Σταματούμε λοιπόν στα 12 χρόνια ηλικία για τα παιδικά προϊόντα. Διευκρινίζει ποιο είναι ο ορισμό αυτό σχετικά με το χρώμα που χρησιμοποιείται, με την περιεκτικότητα σε μόλιβδο και ούτε καθεξής. Εξετάζουμε επίσης και τα προϊόντα που έχουν σχέση με την φροντίδα των παιδιών. Γνωρίζετε ότι χρησιμοποιούνται χημικά με διαφορετικούς τρόπους. Και ένας τρόπος είναι ε, τα χρησιμοποιούμε στα πλαστικά για να είναι πιο ευέλικτα. Ε, υπάρχουν και στους παιδικούς σταθμούς, ε, στα παιχνίδια, σε διάφορα άλλα παιδικά ε, αντικείμενα για παιδιά και δουλεύουμε σε αυτό το νέο ορισμό, ούτω ώστε οι κατασκευαστές και οι καταναλωτές να γνωρίζουν τι καλύπτει ο νέος κανόνας. Επίσης καθορίζει, θα προσδιορίσουμε μάλλον τη λέξη παιχνίδι. Μπορεί να θεωρήσει ότι είναι απλό, αλλά μερικές φορές είναι κάτι που πιο περίπλοκο. Ε, θα είναι ε, οποιοδήποτε αντικείμενο προορίζεται για ένα παιδί νεότερο των 12 ετών. Επίσης, ε, παιδι, ε, αντικείμενα για τη φροντίδα των παιδιών κάτω των τριών ετών. Επίσης, ε, Έχουμε ένα πάνελ από 7 εμπειρογνώμονες ε, για επικίνδυνα αντικείμενα. Έχει δύο διεθνή μέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έναν από το Ηνωμένο Βασίλειο και έναν άλλο επιστήμονα από τη Γερμανία. Ε, θα συνέρθουν φέτος την Άνοιξη και θα συνήλθαν μάλλον και θα κοιτάξουν τις ε, μόνιμες απαγορεύσεις και αν θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, τις απαγορεύσεις αυτές. Επίσης, ένας νέος κανόνας για μια βάση δεδομένων. Θα είναι φιλική προς το χρήστη ε, για... και θα αφορά ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με επικίνδυνα αντικείμενα. Παραδείγματο χάρη, ένα ε, καταναλωτή αγόρασε ένα προϊόν το οποίο δεν λειτουργεί ή προχωρά ή τραυματισμό. Μπορείτε να πάτε σε αυτή τη δημόσια βάση δεδομένων, να έρθετε σε επαφή με, μαζί μας και να μας πείτε ποιο ήταν το πρόβλημα. Με αυτόν τον τρόπο ε, θα πάρουμε πληροφορίες real time ε, πέρα από τις αναφορές που θα που λαμβάνουμε, γιατί μερικές φορές για να φτάσουν ας πούμε, οι, αναφορές χρειάζονται χρόνια. Επίσης, οι κατασκευαστές ε, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια χωριστή πύλη στο διαδίκτυο για τέτοια θέματα. Επίσης, ένα κανόνα για τα τρίτα μέρη που αφορά συγκεκριμένα τους, κατασκευαστές και τις ε, προϋποθέσεις για τις δοκιμές των προϊόντων του, σε περίπτωση που τα προϊόντα αυτά αφορούν τα παιδιά ή δεν αφορούν τα παιδιά. Παραδείγματος χάρη να κατασκευάζετε πούμε, παιχνίδια. Θα πρέπει να δείχνετε ότι έχετε ένα πιστοποιητικό από έναν εξάρτητο ε, εργαστήριο, ότι το, υπήρξε δοκιμή, ότι το δοκιμάσατε ας πούμε αυτό το προϊόν πριν ε, να σας αφήσουμε να το εισάγετε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, για αντικείμενα που δεν αφορούν τα παιδιά, ε, έχουμε πληροφορίες για το πώς ε, θα πρέπει να σέβεστε τα γενικά πρότυπα που αφορούν τα αντικείμενα που δεν απευθύνονται σε παιδιά. Επίσης, ε, τις κούνιες. Μέσα σε νέα χρόνια είχαμε 32 θανάτους και μέσα σε πέντε χρόνια ανακαλέσαμε 7 εκατομμύρια ε, κούνιες γιατί είχαν πρόβλημα. Κάποια παιδιά, κάποια μωρά ε, σφήνωσαν ανάμεσα στο στρωματάκι και στο ε, εξωτερικό ας πούμε της κούνιας και πέθαναν από ασφυξία. Ε, είχαμε πάρα πολλά τέτοια προβλήματα. Το πρότυπο ε, θα ολοκληρωθεί φέτος για τις ε, κούνιες, ε, μέχρι το τέλος δηλαδή, του 2010. Το, το νέο πρότυπο θα μιλάει για το μέγεθος, για τις φορητές κούνιες, όλες οι κούνιες που πουλούνται μέρα μετά την συγκεκριμένη θέση ημερομηνία σε ισχύ με το πρότυπο θα πρέπει να συμμορφούνται με το πρότυπο. Επίσης, το πρότυπο αυτό θα εφαρμοστεί αναδρομικά για κούνιες ε, σε παιδικούς σταθμούς ε, και σε δημόσια μέρη, σε ξενοδοχεία, σε μοντέλ κτλ. Σε οποιοδήποτε μέρος ε, που μπορεί να βρει κανείς κούνιες δημόσιες. We're Επίσης, έχουμε ένα πρότυπο για υποχρεωτική δοκιμή ένα κατασκευαστής ετοιμάζει ένα πιστοποιητικό για να πει ότι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας έχει παράγει ε, ένα αντικείμενο το οποίο δεν ξεπερνάει τις ποσότητες μολύβδου. Παραδείγματο χάρη φτιάξετε μία κούκλα και αγοράσατε ας πούμε ε, τα μάτια από εδώ, τα παπούτσια τα οποία μπορεί να είναι πλαστικά και φτιάξατε την, την κούκλα ε, έτσι συναρμολογώντας την. Αν δείξετε ότι τα επιμέρους ε, τμήματα της κούκλας δεν ξεπερνούν τα πρότυπα, σε, τα όρια μάλλον σε μόλιβδο, τότε δεν χρειάζεται να κάνετε δοκιμές και να ξαναλέξετε ολόκληρη την κούκλα. Αλλά θα πρέπει να έχετε τα πιστοποιητικά από τους κατασκευαστές οι κατασκευαστές θα πρέπει να γνωρίζουν όλη την αλυσίδα των προμηθευτών τους, θα πρέπει να τους εμπιστεύονται και εμείς κάνουμε κάποιες επιτόπιες ε, δοκιμές ή ελέγχους για να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτούς τους ε, προμηθευτές για τις δοκιμές που γίνονται στα επιμέρους τμήματα του αντικειμένου. Επίσης, έχουμε έρθει σε επαφή με όλους τους stakeholders για πρώτη φορά και έχουμε διάλογο επικοδομητικό για να τους ενημερώσουμε για τους νέους κανόνες. Μία από τις προτεραιότητές μου είναι να έρθω σε επαφή α, με αυτούς τους ανθρώπους, να τους εκπαιδεύσουμε, να να παιδαγωγήσουμε για τους νέους κανόνες και κανονισμούς. Ε, το προσωπικό μας κάνει μια τεράστια προσπάθεια διαφορήσης, ούτως ώστε να βοηθήσει τον κόσμο να συμμορφωθεί με τα πρότυπα της Επιτροπής μας. Ε, ο κόσμος ε, έχει ανταποκριθεί με ένα εντυπωσιακό τρόπο. Έχουμε κάνει πάρα πολλά εργαστήρια και έτσι, συνεδριάσεις. Ε, μία τέτοια διάσκεψη κράτησε δύο μέρες και είχαμε 250 ε, συμμετέχοντες. Κάναμε πάρα πολλές επίσης, εκατοντάδες στο ίντερνετ για να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους που έχουν νέες ευθύνες υπό τον νέο νόμο στην σημερινή παγκόσμια αγορά πιστεύω ότι είναι απαραίτητο η Επιτροπή μας να εκπαιδεύσει τον κόσμο όχι μόνο στην Αμερική αλλά και στο εξωτερικό, όχι μόνο τους Αμερικανούς κατασκευαστές της κυβερνήσης, τους καταναλωτές και τους εισαγωγείς, ούτως ώστε τα προϊόντα να είναι ασφαλή. Επίσης κάνουμε ερχόμαστε σε επαφή με ξένες κυβερνήσεις για να προωθήσουμε την κατάρτιση, αλλά θα κάνουμε και άλλες προσπάθειες. Κάνουμε ενημέρωση για κυβερνήσεις, για κατασκευαστές, πολύ τακτικά, αλλά συνειδητοποιούμε ότι θα πρέπει να φτάσουμε και σε χώρες, άλλες χώρες, να φέρουμε τους αξιωματούχους των κυβερνήσεων στις ΗΠΑ για να τους ε, εκπαιδεύσουμε τόσο να καταλάβουν τι θέλουμε. Ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές είναι να δώσουμε τη μάχη ε, πραγματικά στην πρώτη γραμμή του πυρός. να φτιάξουμε δηλαδή ασφαλή προϊόντα, να μην ξοδέψουν εκατομμύρια ε, δολάρια οι κατασκευαστές για να φτιάξουν προϊόντα τα οποία δεν είναι ασφαλή. Θα είμαστε λοιπόν πιο ε, Άγρυπνη σε επίπεδο πρόληψης. Και θα έχουμε ένα τέτοιο νέο γραφείο για αυτές τις επαφές. Επίσης, θα συνεργαστούμε με τους διεθνείς μας εταίρους για περισσότερη κατάρτιση και ελπίζουμε να διοργανώσουμε περισσότερα σεμινάρια, ούτω ώστε μαζί με άλλους εταίρους όπως με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προωθήσουμε αυτή την εκπαιδευτική προσπάθεια. Δεν θα ταξιδέψουμε στο Βιετνάμ, αλλά ξέρουμε ότι εκεί οι άνθρωποι θέλουν να συμμορφωθούν, θέλουν να μάθουν τι, θέλ, τι απαιτούμε. Μας λένε, ε, πέστε μας τι απαιτείτε από μας. Εγώ θα με επωφεληθώ από αυτή την ε, επιθυμία να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια ήδη ε, σε όλη την αλυσίδα κατασκευής ενός ε, αντικειμένου. Νομίζω ότι είναι καλό και για τη χώρα μου και για όλες τις χώρες όπου εισάγονται πάρα πολλά προϊόντα. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητές μου, αυτή η συνεργασία. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά ακόμα, να σας ε, μιλήσω για τις παρελθούσες και τις σημερινές δραστηριότητες της ε, Επιτροπής μας. Εμείς έχουμε 50 νέους κανόνες, ε, έγγραφα, κατευθυντήριες γραμμές, εφαρμόσουμε δηλαδή σε όλα τα μέτωπα τον νέο νόμο. Επίσης το, προσωπικό μας, το προσωπικό μας ε, έρχεται σε επαφή με τους stakeholders για να τους ενημερώσει για τις προϋποθέσεις και συνεχεία προσπαθεί να τους εκπαιδεύσει για το πώς θα συμμορφωθούν. Κινούμαστε με ταχύτητα τους ρυθμούς ε, και είμαι πολύ περήφανη που είμαι επικεφαλής αυτής της προσπάθειας. Όπως βλέπετε στην Επιτροπή έχουμε ανασκουμπωθεί πραγματικά, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ε, εστιαζόμαστε κυρίως στο σημαντικούς νέους ορισμούς ε, που εντάσσουν διάφορες ασφαλιστικές ε, δικλίδες στην όλη προσπάθεια, ούτως ώστε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Επίσης, ε, θέλουμε να έχουμε πιο στενές επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μπορούμε να μιλάμε όπου γίνεται με ενιαία φωνή. Μια κοινή αποστολή είναι τα προϊόντα να σχεδιάζονται με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, να πιστοποιούνται από πιστοποιημένα εργαστήρια και να μην προκαλούν τραυματισμούς. Υπάρχει μία δέσμευση για την ασφάλεια αυτών που υπηρετούμε. Αυτή πρέπει να είναι η κοινή μας αποστολή. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να έρθω εδώ και να σας μιλήσω. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Πιστεύω ότι έχουμε κάποιες θεμελιώδεις αρχές που μας, κάνουν, που μας επιτρέπουν να συνεργαστούμε και πραγματικά θέλω να συνομιλήσω μαζί σας για να ανταλλάξουμε πληροφορίες για τις κοινέ μας δραστηριότητε. Με χαρά θα απαντήσω στις ερωτήσεις. Well, thank you very much indeed. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αλλά και ενθαρρυντική η ε, παρέμβασή σας. Πραγματικά εντυπωσιάζομαι από τι εξελίξει Έχω συναντήσει παλαιότερα, έχω γνωρίσει την προκάτοχό σα. Και αυτό που είπατε στην αρχή, δηλαδή ότι χρειάζεται μια αγορά με ανθρώπινο πρόσωπο, Ακριβώ βρίσκεται στο επίκεντρο και του δικού μα ενδιαφέροντος. Και πρόσφατα περάσαμε μια, κλείναμε μια έκθεση του κ. Γκρέκ εδώ, συναδέλφου μας, ε, για μια κοινή αγορά πολιτών και καταναλωτών. Και αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό για μας. Νομίζω ότι έχουμε πράγματι ένα μεγάλο σύνολο θεμάτων και πολλοί συναδελφοί μου θα θελήσουν να παρέμβουν. Θα παρακαλέσω όμως πρώτα τον κύριο Μορέρα να μιλήσει και μετά ο κύριος Κρότσμαν που αντιμετωπίζει πίεση χρόνου θα λάβει το λόγο και μετά θα ακούσω τους άλλους συναδέλφους. Αλλά έχουμε και νέο βουλευτή, την κυρία Σάντια Λούβα. Πολύ ευχαρίστως να λάβετε το λόγο αργότερα αν θέλετε. Και που γνωρίζω ότι είναι και μέλη από την ε, Επιτροπή Προστασίας Υγείας και Καταναλωτών. Τώρα, ας ακούσουμε τρεις-τρεις τους ερωτώντες. Πρώτα όμως ο κύριος Ευχαριστώ και συγχαίρω την Επιτροπή σας για την οργάνωση της ε, παρούσας συνεδρίασης που νομίζω ότι είναι και επίκαιρη και θα αποδειχθεί και καρποφόρα. Η παρουσίαση της Προέδρου ε, της Επιτροπής ε, Ασφάλειας Προϊόντων Καταναλωτού είναι σημαντική διότι γνωρίζουμε τις βελτιώσεις που έχουν επέλθει στο ρυθμιστικό πεδίο, στο νομοθετικό και ρυθμιστικό πεδίο για την προστασία των καταναλωτών στις ΗΠΑ Και επειδή και εμείς είμαστε υπερήφανοι για τις δικές μας προδιαγραφές, Χαίρομαι που βλέπω οι Ηνωμένε Πολιτείε να συγκλίνουν μαζί μας για θέματα προστασίας και ασφάλειας των προϊόντων γιατί μαζί η επιρροή που μπορούμε να ασκήσουμε στην παγκόσμια οικονομία μπορεί να μας κάνει να είμαστε πρωτοπόροι και για την προστασία των καταναλωτών αλλά και για το παγκόσμιο εμπόριο. Και αυτή είναι μια πτυχή που θα ήθελα να επισημάνω και να τονίσω την σημασία των ρυθμιστικών πτυχών όχι μόνο στο διμερές εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, αλλά και στο παγκόσμιο εμπόριο, γιατί όπως γνωρίζετε, τα κολλήματα στο εμπόριο δεν είναι μοναχά δασμολογικά. Υπάρχουν και οι διαφορές στην νομοθεσία, στις ρυθμίσεις και ιδιαίτερα στις προδιαγραφές ασφαλείας των προϊόντων που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κόλλημα στις ε, συναλλαγές. Ως γνωρίζετε έχουμε ε, γερά θεμελιωμένες πλέον ε, σχέσεις με, ε, τις, με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αλλά μπορούν να βελτιωθούν έτσι περαιτέρω. Και ένας τρόπος θα ήταν να εναρμονιστούν οι προδιαγραφές ασφαλείας. Και βλέπουμε πολύ καλό μάτι αυτή τη συνεργασία μεταξύ ημών αφενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκών Θεσμών και των Ενωμένων Πολιτειών, των αντίστοιχων θεσμών των Ενωμένων Πολιτειών. Και θα αποβεί νομίζω κρίσιμο αυτό, η κρίσιμη προσπάθεια αυτή για την κατάργηση ή μείωση τουλάχιστον όσο είναι δυνατόν των φραγμών στο εμπόριο. Εάν μπορέσουμε δηλαδή να εναρμονίσουμε σε υψηλό βέβαια επίπεδο τις προδιαγραφές μας, αν λοιπόν καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, θα μπορέσουμε να απαλείψουμε ορισμένα από τα πιο σημαντικά κολλήματα στο εμπόριο. Η άλλη πτυχή είναι το παγκόσμιο εμπόριο. Εάν οι δύο πλευρές μας συνεννοηθούν για τις προδιαγραφές. Μπορούμε έτσι να καταδείξουμε στους άλλους σημαντικούς εταίρους για παράδειγμα ε, κατασκευαστές παιχνιδιών, οικιακών συσκευών, ότι είναι κρίσιμο για την επιβίωσή τους να συμμορφωθούν με τις προδιαθέσεις ασφαλείας των ΗΠΑ και της ΕΕ. Άρα πάλι θα εκπληρώσουμε έτσι σημαντική αποστολή σε ό,τι αφορά την διευκόλυνση της, ε, του παγκόσμιου εμπορίου, που είναι σημαντικό για την δημιουργία απασχόληση και για το παγκόσμιο εμπόριο. Έτσι λοιπόν, ως Πρόεδρος Επιτροπής, άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εισήγησή σα, κυρία Πρόεδρε για την ασφάλεια των προϊόντων στις ΗΠΑ. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα την συνεισφορά που μπορούμε να κάνουμε οι δύο πλευρές του Ατλαντικού για να βελτιωθούν οι συνθήκες όπως είπα για να βελτιώσουμε τις ήδη καλές σχέσεις που έχουμε και στις επενδύσεις αλλά και για την καθιέρωση κοινών προδιαγραφών τις οποίες να σέβονται και άλλοι σημαντικοί παραγωγή Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ πολύ για την συνεισφορά σας στη συζήτηση. Πρόεδρε, εμείς υποστηρίζουμε πάρα πολύ την εναρμόνιση των προδιαγραφών και των προτύπων. Και επίσης, ελπίζουμε ε, να ε, δράσουμε από κοινού με την Ευρώπη και τον Καναδά ε, για να έρθουμε σε επαφή με κατασκευαστές ε, παραθύρων ε, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στα ρολάκια της γρίλες και τα παιδιά μπλέκονται στο λουρί που ανοίγει και στραγγαλίζονται. Γιατί υπάρχει αυτή η φιλιά ε, και ε, μπορούν να κατασκευαστούν ρολά ας πούμε και ε, χωρίς καθόλου ταινία λουρί. Μπορούμε λοιπόν να δούμε ποιε είναι οι προδιαγραφέ, ποια είναι τα πρότυπα που να βασίζονται όμω σε επιστημονικέ ε, ανακαλύψει και στοιχεία και να ε, συνεννοούμαστε με τον Καναδά και την Ευρώπη, οι Ηνωμένε Πολιτείε, για να επηρεάσουμε και του κατασκευαστέ και να υιοθετούν τι βέστιστες ε, πρακτικέ και εμείς θέλουμε βεβαίως να ε, είναι ασφαλείς οι καταναλωτές μας, αλλά και οι προδιαγραφές των παιχνιδιών μας δεν ε, επηρέασαν το εμπόριο με την Κίνα. Κάθε χρόνο ο αριθμός των καταναλωτικών προϊόντων, ο συνολικός εννοώ, ε, των εξαγών από την Κίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζει να αυξάνεται. Είμαστε από τους μεγαλύτερους καταναλωτές κινέζικων προϊόντων. Ε, αυτό δεν τους έχει επηρεάσει λοιπόν το γεγονός ότι έχουμε ψηλά πρότυπα ασφαλείας για παιχνίδια και άλλα προϊόντα που εισάγουμε. Δεν το θεωρούμε καθόλου φραγμό. Μάλλον ε, καλή πρακτική για προστασία των καταναλωτών. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μία ερώτηση μόνο έχω. Είπατε ότι οι εταιρείε που φέρουν τα προϊόντα του στην αγορά σα θα πρέπει να έχουν ε, πιστοποίηση. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η υποπτία των αγορών. Γιατί ε, ωραίε είναι οι προδιαγραφές και πολύ ενδιαφέρον να δηλώνει κανείς ότι τη στηρεί. Αν δεν υπάρχει όμως λειτουργούσα υποπτία της αγοράς και έλεγχο κυκλοφορούν μεν τα προϊόντα και αναφέρει ότι ε, χρησιμοποιεί τα πιο σύγχρονα προϊόντα και όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κάποια κενά γιατί τα κράτη-μέλη παραμένουν ε, αρμόδια για τον έλεγχο της αγοράς και έχουν διαφορετικές ε, προδιαγραφές. Ας πούμε ότι αυτά είναι τα προϊόντα σε ένα λιμένα. Τι γίνεται, πώς τα ελέγχετε, αν είναι στις προδιαγραφές σας ή όχι. Αυτό πώς ε, εξακριβώνεται. Θα με ενδιαφέρει. Thank If you manufacture a children's toy or uh, if you're domestic manufacturer. Λοιπόν, για τα παιχνίδια. Όταν είναι κάποιο ε, εισαγωγέα και όχι μόνο παιχνιδιών, γενικά για προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά, θα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό από εργαστήριο που να ε, διαβεβαιώνει ότι ε, συμμορφούνται προς την νομοθεσία και δεν ε, υπερλαμβάνει ε, ε, μόλιβδο περισσότερο από όσο πρέπει ή φθαλικές ενώσεις περισσότερες από όσο πρέπει στο και καθόλου. Και θα πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο πιστοποιητικό. Δεν μπορούν να εκφορτωθούν λοιπόν στι ΗΠΑ τα προϊόντα, δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά αυτά και τα πιστοποιητικά. Αυτός είναι ένας τρόπος, ο έλεγχος το λιμένα. Ένας άλλος τρόπος είναι ότι πηγαίνουμε στα καταστήματα, αγοράζουμε τα προϊόντα, στα ράφια και τα ελέγχουμε. Έτσι. Επίσης, οργανώσεις καταναλωτών και ε, δικηγόροι καταναλωτών αγοράζουν προϊόντα. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα τέτοιο ε, επεισόδιο με γυαλιά. Καλή είναι η υποπτή όμως περίχαν κάδμια. Έχει αλλάξει λοιπόν η δυναμική της αγοράς με την καινούργια νομοθεσία. Για παράδειγμα, στην Κίνα, εκείνοι που παράγουν φερμοάρ ή κουμπιά, ε, θα πρέπει να δουν ε, ότι ε, φτιάχνουν προϊόντα που, δεν, που είναι ελεύθερα μολύβδου και φθαλικών ενώσεων και τα φερμοάρ και τα κουμπιά. Λοιπόν, αλλάζουμε τη δυναμική της αγοράς, γιατί αν κάποιος θέλει να πουλήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 90 ppm ε, ε, σε μολύβδο και 300 ppm σε ενώσεις μολύβδου. Γίνεται λοιπόν έλεγχος και επιστοποίηση και αυτό είναι ένα εργαλείο ε, εφαρμογής του νόμου για να μην μπαίνουν ε, τέτοια προϊόντα στην Αμερικανική αγορά. Ξέρω ότι υπάρχουν και απομιμήσεις βέβαια και των πιστοποιητικών, το γνωρίζουμε αυτό και επαγρυπνούμε. Και επίσης ζητούμε από τους κατασκευαστές όχι μόνο να επιδεικνύουν αυτά τα πιστοποιητικά, αλλά να έχουν και ένα ε, έτσι, λογικό πρόγραμμα ελέγχου όταν αλλάζουν τα υλικά, να το ξαναελέγχουν αλλά να ελέγχουν και τα εργαστήρια σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ε, είναι σίγουροι ότι είναι σωστά και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, έχουμε αυτό το σύστημα ε, απαιτήσει ελέγχου και επιστοποίηση και αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό του μολύβδου και των φθαλικών ενώσεων και ζητούμε και από τους κατασκευαστές και όταν χρησιμοποιούν κάποια εξαρτήματα, κάποια ανταλλακτικά, ε, να παρακολουθεί τη αλυσίδα μέχρι τον κατασκευαστή για να μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι είναι γνήσια τα πιστοποιητικά υψηλή ποιότητα στα εργαστήρια και να του εμπιστευόμαστε. Δεν μπορεί κανένα εργαστήριο να ελέγξει και να δώσει πιστοποιητικό εάν δεν το έχουμε εγκρίνει εμείς. Είναι εγκεκριμένα πιστοποιημένα και τα ίδια τα διαπιστευμένα μάλλον τα εργαστήρια. Ότι έχουν τη δυνατότητα και το έχουμε εμείς αναγνωρίσει και το δηλώνουμε ότι είναι σε θέση μάλιστα να ελέγχουν σωστά ε, τα προϊόντα. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα επίπεδα ασφαλείας και βαθμίδες. Είναι περίπλοκο, δεν ξέρω. Α, θα ήθελα να σας συστήσω και το Ρίτσαρντ Μπράιαν. Ο Ρίτσαρντ Μπράιαν είναι ο Διευθυντής ε, των Διεθνών ε, Υποθέσεων στην Επιτροπή μας και πολλά χρόνια έχει εργαστεί στην εξωτερική υπηρεσία, συνεργάζεται με την Κίνα και χρόνια ολόκληρα με κατασκευιστέ. Και είναι εδώ και ο Ματ Χάουσερ, ο προσωπάρχης μου και ε, νομικός μου σύμβουλος και αν ε, νομίζει ότι είναι σκόπινο να μιλήσει μπορεί να πάρει το λόγο ή να μου δώσει κανένα σημείωμα να τα πω εγώ. Μάλιστα. Με μεγάλη χαρά θα του δώσουμε το λόγο. Θέλω να σας πω ποιοι συνάδελφοι τώρα θα ε, κάνουν ερωτήσεις η κυρία Σάλντε Μόζερ και μετά προηγουμένω σα τη συνέστησα κυρία Τενμπάουμ να πω και στους υπολείπους ότι ορίστηκε η συγγήτρια της Επιτροπής μας στην έκθεση που κάνουμε για την αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων. Θα δούμε τι πολιτική και τι στρατηγική θα ακολουθήσουμε και πραγματικά ενδιαφέρει το θέμα. Η κυρία Βανιού, η κυρία Τούν και η κυρία Τάιλερ. Αν θέλει και κανένας άλλος, παρακαλώ ζητήστε το λόγο. Και ο καθηγητής Κορέντε Κάμπος, αν θέλει αργότερα. Η κυρία Σάλντε Μόζερ πρώτη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας, κυρία Τένενμπαουμ. Πολύ χρήσιμο και πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον για μένα, στη δική μου δουλειά. Έχω ε, και πολλές ερωτήσεις να σας κάνω, δεν θα τις θέσω όλες τώρα. Πρώτον, έχετε δει ήδη από τώρα μείωση ε, στους τραυματισμούς και τα ατυχήματα μετά από το νέο αυτό καθεστώς. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το μάθουμε. Μιλήσατε επίσης για εχνηλασιμότητα των προϊόντων. Αυτό μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε. Πώς ε, είστε βέβαιοι ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε πάντα την προέλευση. Και θα ήθελα ε, να δω πώς ε, θέτεται και τα πρότυπα και τις προδιαγραφές στις Ηνωμένες Πολιτείες με εκπροσώπους των εταιριών, των καταναλωτών, των κρατικών αρχών. Ποιος συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια ορισμού των προδιαγραφών και των προτύπων. Και ένα τελευταίο. Έχετε διαφορετική μεταχείριση ε, ανάλογα με τις πωλήσει, αν είναι διαδικτυακές ή στην αγορά, γιατί θα μιλήσουμε εδώ για τον DPST στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Thank you. Uh, ευχαριστώ, κυρία Σκάλντε Μόζε, για τις ερωτήσεις σας. Υπήρξε δραματική μείωση στις ανακλήσεις προϊόντων, ε, ειδικά για λόγους μολύβδου. Όλα τα στοιχεία μας ε, μπορείτε να τα βρείτε στο, στην ιστοσελίδα cpsc.gov. Υπάρχει μείωση λοιπόν στις ανακλήσεις. Δεν έχω τα δεδομένα μαζί μου, αλλά ελπίζω με αυτόν τον τρόπο ε, να έχουμε και μειώσεις ε, στις επαφές ε, των παιδιών με μόλιδο που, που δημιουργεί πρόβλημα στον εγκέφαλο. Επίσης, η ανιχνευσιμότητα είναι πολύ σημαντικό ε, η φιλαλήθεια των πιστοποιητικών για τα εξαρτήματα. Για να είμαστε σίγουροι, για να είναι σίγουρος ένα κατασκευαστής, θα πρέπει να γνωρίζει τους προμηθευτές του και θα πρέπει περιοδικά να ελέγχονται οι προμηθευτές του, ώστε να μπορεί να βασίζεται στους προμηθευτές ε, για τα εξαρτήματα. Ε, υπάρχει λοιπόν αυτή η ανιχνευσιμότητα. Τώρα υπάρχει και η νεοτεχνολογία στην διάθεσή μας. που μαζί με διάφορους ομοσπονδιακούς φορείς και εταίρους για την έρευνα στην ε, νανοτεχνολογία, ούτω ώστε να ξέρουμε τι συμβαίνει, γιατί ο τομέας αυτός ε, εξελίσσεται ταχύτατα και θέλουμε να υπάρχει η ανιχνευσιμότητα των νανοηλικών. Επίσης θέλουμε μία ετικέτα προέλευσης των παιδικών παιχνιδιών και προϊόντων. Θέλουμε το προϊόν να φέρει αυτή την ετικέτα, ούτω ώστε ο καταναλωτής να ξέρει από ποια εταιρεία προέρχεται και από ποια χώρα προέλευσης προέρχεται, που βρίσκεται ο κατασκευαστής. Ανάλογα με το προϊόν, λοιπόν, χρησιμοποιούμε απλώς την κοινή λογική για να δημιουργήσουμε την καλύτερη δυνατή ετικέτα. Έχουμε τους, τους γραμμικούς κωδικούς, έχουμε αυτές τις ετικέτες. Κάποια στιγμή αυτά τα μέσα θα εξαπλωθούν παγκόσμια. Θα έχουμε την, τις πληροφορίες για τα υλικά, την χώρα, την παρτίδα και πολλά από αυτά θα τα βλέπουμε αμέσως ανάλογα με το είδος του κώδικα. Η τεχνολογία λοιπόν εξελίσσεται. Επίσης ε, θα έχουμε και μια στήλη για προϊόντα που ανακαλούνται. Πώς κατασκευάζουμε τα πρότυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Επιτροπή για την Ασφάλεια των Κατανοητικών Προϊόντων επιφορτίστηκε όταν δημιουργήθηκε με τη δημιουργία εθελοντικών προτύπων. Ε, βασιζόμαστε σε φορείς που δημιουργούν τέτοια θελοντικά πρότυπα. ούτω ώστε να, να χρησιμοποιεί αυτά τα πρότυπα η βιομηχανία. Και αν δεν είναι αρκετά στεναρά για να προστατεύσουν το καταναλωτή αυτά τα πρότυπα, τότε μπορούμε να περάσουμε σε υποχρεωτικά πρότυπα. Για τα προϊόντα τα παιδικά είδαμε ότι τα πρότυπα αυτά ε, δεν ήταν αρκετά αυστηρά για να μας να προστατεύσουν ας πούμε, ε, για τις βρεφικές κούνιες, ε, για τα καρεκλάκια, τα καθισματάκια κτλ. Και για τα παιχνίδια επίσης ε, θα τα καταστήσουμε πιο αυστηρά τα πρότυπα. Ένας τρόπος λοιπόν με τα πρότυπα, όπως κάνουμε με τις βρεφικές κούνιες, δουλεύουμε το ISTM, το φορέα αυτό, του λέμε τι θέλουμε, Υπάρχει ένα νέο πρότυπο και μάλιστα φέτος ε, θα περάσουμε ένα νέο πρότυπο, ούτως ώστε να μην, να, πουλά, να μπορεί να πουλήσει βρεφικές ε, κούνιες που έχει ένα τμήμα, πούμε, το οποίο είναι πτυσσόμενο και ανοίγει και κλείνει. Επίσης θέλουμε καλύτερα υλικά, γιατί καμιά φορά το πλαστικό έφευγε από το ξύλο και τα παιδιά πεθαίνουν από ασφυξία γιατί όταν αποκολλάται πούμε το πλαστικό από το ξύλο, τα παιδιά σφινώνονται ε, ανάμεσα και πέθανε από ασφυξία. Δουλεύουμε με το STM, ε, το φορέα αυτό, ε, του είπαμε τι ακριβώς θέλουμε, υιοθέτησαν τις, α, τις απαιτήσεις μας. Δουλεύουμε δηλαδή με το φορέα, φτάνουμε σε μια συνένεση, φτάνουμε, φτιάχνουμε το υψηλότερο δυνατό ε, πρότυπο και το επιβάλλουμε υποχρεωτικά. Κάτι άλλο που κάνουμε, ε, κάνουμε έρευνα. Χρησιμοποιούμε την έρευνα που έχουν κάνει, παραδείγματο χάρη, οι ερευνητέ και οι επιστήμονε σε άλλε χώρε. Κοιτάμε τα δικά σα, περιπεί. Και τότε κάνουμε μια δημόσια συζήτηση, λέμε. Να, εμεί την προτείνουμε. Μπορούμε να ανακοινώσουμε, ας πούμε, ότι θα επιβάλλουμε ένα νέο πρότυπο, ένα νέο κανόνο. Ε, το δημοσιεύουμε, ε, αυτό που προτείνουμε εμείς, ε, για να το σχολιάσει ο κόσμος. Το συζητάμε και μετά αποφασίζουμε α, τελικά πώς θα διαμορφωθεί. Επίσης το Κογκρέσο. Μιλάει για, νομοθετικά ας πούμε, αποφασίζει για τον α, ε, μόλιδο, παραδείγματος χάρη, 90 ppm 90 στα 1000. Ε, του χρόνου θα γίνει 100. στο εκατομμύριο, συγγνώμη. Έχουμε προσωπικό στο CPSC επίσης που κοιτάει το eBay και και υπάρχει μια ενημέρωση ε, του eBay, ας πούμε, ε, για τις ανακλήσεις προϊόντων. λέμε, ας πούμε, δεν μπορεί να πουλήσετε αυτά τα προϊόντα. Επίσης, ε, για τις ε, δημοπρασίες που γίνονται, Φερρυπίν στην Ατλάντα, στην, στη Γεωργία. πάμε εκεί, στέλνουμε προσωπικό και ενημερώνουμε για τα προϊόντα. Είμαστε μικρή υπηρεσία, αλλά είμαστε πολύ δραστήρια. Έχουμε κάτι παραπάνω από 500 υπαλλήλου για όλες τι ΗΠΑ. Δεν είμαστε μεγάλη υπηρεσία. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Όταν, όταν δεν έχει κανείς πολύ προσωπικό, πρέπει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία. Πρέπει να καταφύγει σε αυτό το μέσο. Και αν μια εταιρεία δεν συμμορφωθεί ε, με τους κανόνες σας. Υπάρχουν, να προβλέπονται κυρώσεις, ποιες είναι οι επιπτώσεις. Ναι, έχουμε και αστικές και ποινικέ κυρώσεις. Το 2008 επιβάλαμε τις ποινικέ κυρώσεις. Μπορούμε να επιβάλλουμε πρόστιμα, μπορούμε να τους πούμε ότι αποκλείονται από την Αμερικανική αγορά. Μια εταιρεία, Dezo λέγεται, Ε, η οποία αγνοούσε τους κανόνες μας, ε, της επιβλήθηκε ένα τεράστιο πρόστιμο. Και έχουμε ένα σχέδιο ολόκληρο που θα τις επιβάλλουμε, ούτως ώστε να μην να, ε, μας αγνοεί. Μπορούμε να κάνουμε και ποινική δίωξη, αλλά κάποια στιγμή σταματάει η εμπορική τους δραστηριότητα, αν μας αγνοούν. fine. Το πρόστιμο μπορεί να φτάσει στα 15 εκατομμύρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρήσιμο και το υλικό αυτό για την έκθεση της Κρίστελ νομίζω. Η κυρία Βαρνιό που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω κυρία Τένενμπαουμ ε, για την παρουσία σας ενώπιον μας. Είχα διαβάσει το βιογραφικό σας και με εντυπωσίασε ιδιαίτερα ε, το έργο σας όλα αυτά τα χρόνια και ε, το αποτέλεσμα. Σε λίγο κλείνεται ένα μόλις χρόνο στη θέση αυτή και έχετε κάνει τόση δουλειά. Μιλήσατε για πρότυπα και προδιαγραφέ, ε, υποχρεωτική εφαρμογή και σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Θέλω να σα κάνω μερικέ ερωτήσει. Μιλήσατε για εκπαίδευση, για κατάρτιση και ενημέρωση του προσωπικού μέσω εργαστηρίων. Πολύ ε, ουσιώδης και θεμελιώδης αυτό μου φαίνεται για την προστασία των καταναλωτών. Γιατί θα πρέπει να συμμετέχουν και οι πολίτες ενεργά στην προστασία των καταναλωτών. Θέλω λοιπόν να σας κάνω την εξής ερώτηση. Πώς μπορείτε να συνεργάζεστε με ε, οργανώσεις καταναλωτών ε, για να ε, ενημερώνουν τους καταναλωτές και τι ποσοστό του προπολογισμού σας αφιερώνεται σε αυτή την προσπάθεια. Μιλήσατε επίσης για σεμινάρια, για ενίσχυσή τους, σεμινάρια μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά για τη συνεργασία για να έχουμε κοινά στάνταρ, κοινέ προδιαγραφές και να μπορούμε καλύτερα να επηρεάζουμε ε, τις ε, πρακτικές των εταιριών παγκοσμίω. Θέλω να σας κάνω την εξερώτηση. Πολύ μεγάλη φιλοδοξία και μπράβο σας. Είναι πολύ ωραίο να έχει κανείς τόσο υψηλές φιλοδοξίες. Πιστεύετε όμως ότι μπορεί κανείς γρήγορα να προχωρήσει ε, συνεργαζόμενος Δηλαδή εμείς με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταπολεμήσουμε και τις απομιμήσεις και μέσω του διαδικτύου, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το εξή πρόβλημα. Έχουμε διαφορετικέ προδιαγραφέ στα διάφορα κράτη μέλη, 27 κράτη, και δεν είναι πάντα το ίδιο επίπεδο ε, τη ενημέρωση και τη εκπαίδευση και τη κατάρτιση και τη γνώση των καταναλωτών και των ε, οργανώσεών του. Και στα θεσμικά όργανα η προστασία του καταναλωτού είναι σε διάφορες ε, επιτροπές και σε διάφορους επιτρόπους. Δηλαδή, έχετε μήπως κανένα πρόβλημα ποιο να πάρετε τηλέφωνο στην Ευρώπη, σε ποιο να αποταθείτε. Θα θυμάστε τι είχε πει κάποιος, ότι δεν θέλω να μιλήσω με την Ευρώπη, ποιο να πάρω το στο τηλέφωνο. Thank you. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσεις για να δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια σε ό,τι με αφορά προσωπικά. Με τον προϋπολογισμό που διαθέτουμε στα εργαστήρια και στην ε, εκπαίδευση. 118 εκατομμύρια ε, έχουμε το χρόνο. 118 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Για όλο τον οργανισμό δεν είναι πολλά χρήματα. Για ένα μικρό ποσοστό πηγαίνει στην εκπαίδευση και στη διάδοση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη συνεργασία με άλλους για να μπορούμε να φτάνουμε ε, στους τελικούς αποδέκτες για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των καταναλωτών. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να συμμετέχουμε και στον ΩΣΑ αλλά και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεργαζόμαστε με το κέντρο αναφοράς και ελέγχου νοσημάτων ε, που και αυτό έχει ως στόχο την πρόληψη ε, ατυχημάτων, τραυματισμών, θανάτων από προϊόντα. Και επίση είναι σημαντικό να συνεργαζόμαστε με πανεπιστήμια, κολέγια και άλλους ομοσπονδιακούς οργανισμούς ε, που επιζητούν τη συνεργασία μας και με διεθνείς ε, φορείς. Γιατί και είναι λογική, δεν είναι, να θέλει κανείς να είναι ενημερωμένος ο πολίτης, ο καταναλωτής, ε, να υπάρχει διάδοση της γνώσης και της ενημέρωσης. Για να ε, δίνουμε περισσότερη έμφαση στην πρόληψη και να μην αντιδρούμε συνεχώς. Από εκεί θέλουμε να ξεφύγουμε από το στάδιο της αντίδρασης. Όχι, να ε, ενεργούμε δραστήρια και εκ των προτέρων. Με κυβερνήσεις συνεργαζόμαστε. Φέτος μόλις ανοίξαμε γραφείο στο Πεκίνο με έναν και ε, ε ντόπιο εργαζόμενο, προσεχώς προσθεθεί και ένας Αμερικανός, και ε, ε, εδρεύουμε στην ε, πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Οι δύο αυτοί λοιπόν υπάλληλοι θα διευκολύνουν τις επαφές μας, τη συνεννόηση με τις κινέζικες αρχές σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή κινέζικων προϊόντων. Και αυτό θέλουμε να το διευρύνουμε βεβαίω. Κάτι άλλο. Για την εκπαίδευση και πάλι και την ενημέρωση. Βεβαίως συνεργαζόμαστε με ενώσεις καταναλωτών, με την ε, Ομοσπονδία Καταναλωτών, ε, Safe Kids. Υπάρχουν διάφορες, δύο-τρεις πολύ ε, γνωστές και σημαντικές οργανώσεις προστασίας καταναλωτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανταλλάσσουμε ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα και διατηρούμε εξαιρέτες σχέσεις. Και ακριβώς εκεί συνεργαζόμαστε. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη και ευρύτερη συνεργασία. για τις απομιμήσεις. Προηγουμένως μιλούσα εγώ για απομιμήσεις ε, πιστοποιητικών. Όταν κάποιο κατασκευαστή πρέπει να φέρει ένα πιστοποιητικό που λέει ότι εγώ παράγω ε, προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά και ε, έχουν ελεγχθεί και δεν περιέχουν μόλιβδο ή φθαλικές ενώσεις ε, παραπάνω από όσο προβλέπετε. Λοιπόν, ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να καταλάβουμε ότι είναι γνήσιο αυθεντικό το πιστοποιητικό, ότι δεν είναι πλαστό το πιστοποιητικό. Τώρα, η απομίμηση προϊόντων προβλέπεται. λοιπον ζήτημα εμπορικών σημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Εμείς δεν έχουμε τέτοια δικαιοδοσία στις απομιμήσεις των αγαθών. Όταν μιλώ για απομιμήσεις εννοώ πλαστά πιστοποιητικά. Αυτό είναι η δική μας αρμοδιότητα. Ε, να προσέχουμε και να ελέγχουμε. Και ως πρώην εκπαιδευτικό, πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό ακριβώς να εκπαιδεύουμε και να βοηθούμε και τις ε, ξένες κυβερνήσεις, όχι μόνο τους ξένους κατασκευαστές. Και να χρησιμοποιούμε τον προϋπολογισμό μας κάθε χρόνο ε, λίγο και, όλο και περισσότερα χρήματα να δίνουμε σε αυτή την πτυχή της εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Πολύ ωραία ερώτηση. is next. Oops, thank you very much. Um, I am very happy that I... Ευχαριστώ, λέει η κυρία Τούν. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτή τη συνεδρίαση. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία σε αυτόν τον ευρύ τομέα των προτύπων. Γιατί χάρη σε αυτή τη συνεργασία μπορεί να βελτιωθούν τα προϊόντα. Πέρυσι και πριν από δύο χρόνια θυμάμαι ότι είχαμε μια κρίση με κινέζικα παιχνίδια που η Κομισιόν ήθελε να τα στείλει πίσω. Ε, είναι σημαντικό να σταματήσουμε τέτοιου τύπου επικίνδυνη παραγωγή. Ε, παρακολουθείτε και τις πωλήσει των ε, προϊόντων που δεν είναι καινούρια, ε, των, που είναι δεύτερο χέρι ή που, πουλιού, που γίνονται σε παζάρια κτλ. Για να παρακολουθήσετε όλη την αγορά και σε αυτό το επίπεδο, στις όλες τις ΗΠΑ, θέλετε πάρα πολύ κόσμο προφανώς για να παρακολουθήσει όλες αυτές τις δραστηριότητε. Κάτι άλλο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, ασχολείστε και με τρόφιμα, γιατί αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Δεν ξέρω καν αν έχουμε το χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Α, δεν ασχολείστε με τρόφιμα. Μου γνέφεται αρνητικά. Επίση, μιλήσατε πάρα πολύ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, συμφωνώ απόλυτα, αυτό το θέμα. Στην κατάρτιση αυτό, είναι, αυτό που είναι σημαντικό είναι να εκπαιδεύσουμε και να καταρτήσουμε αυτούς που παράγουν αυτά τα αντικείμενα και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ένας από τους στόχους σας είναι να υπάρξει συνεργασία για κοινά πρότυπα. Ακόμη πόρο απέχουμε από τα κοινά πρότυπα. Δεν έχουμε καν κοινά πρότυπα εμείς 27 χώρες στην Ευρώπη. Αλλά αν εκπαιδεύσουμε τον τον κόσμο, για τον τρόπο που παράγει, α, ίσως θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό παρανομαστή για τον τρόπο παραγωγής. Και έπειτα, έχετε κανένα παράδειγμα θεαματικής επιτυχίας χάρη στην κατάρτιση, που, σε σεμινάρια κατάρτισης ας πούμε που διοργανώσατε. Μπορείτε να μας δώσετε έτσι ένα παράδειγμα πιο χειροπιαστό. Γιατί πιστεύω ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ε, είναι πολύ επωφελής για όλους τους ενδιαφερόμενους. Ευχαριστώ. Έχουμε κάτι παραπάνω από 500 υπαλλήλου σε όλη την Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων για όλες τις Πολιτείες. Έχουμε 14 αεροδρόμια, του χρόνου θα καλύψουμε 19. Ε, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά με τις θελονιακές αρχές και τις συνοριακές αρχές. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ε, ε, εξυγχρονίζουμε το δικό μας ε, σύστημα μηχανοργάνωσης, ούτως ώστε να εντοπίζουμε τα προβληματικά προϊόντα. Έχουμε μια δημόσια βάση δεδομένων, όπου οι καταναλωτές μπορούν να μας πούνε αν έχουν τραυματιστεί από κάποιο προϊόν. Για να επεκτείνουμε λοιπόν ε, τις δραστηριότητε μας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία. Είναι σημαντικό να συνεργαστούμε και στις ΗΠΑ αλλά και διεθνώς και η συνεργασία θα πρέπει να γίνει και με άλλε ομοσπονδιακέ ε, υπηρεσίες. Εμείς, ας πούμε, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τρόφιμα. Η FDA, η υπηρεσία για τα τρόφιμα, είναι υπεύθυνη. Για τα καλλιντικά, για τα τρόφιμα, για μια σειρά από άλλα προϊόντα. Υπάρχουν άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, άρα η συνεργασία είναι πολύ σημαντική. Τώρα, για αυτό που με, ρωτήσε, με ρώτησε μια βουλευτής... Ε, σε ποιον τηλεφωνούμε. Έχουμε επαφή στη Γενική Διεύθυνση ε, ΣΑΝΚΟ. Έχουμε επαφή με διάφορους φορείς ανά τον κόσμο. Ε, δουλεύουμε και συνεργαζόμαστε με τις πρεσβείες μας και αν έχουμε κάποιο πρόβλημα ερχόμαστε σε επαφή με αυτές τις πρεσβείες και όντως μας βοηθούν. Η συνεργασία είναι η λέξη κλειδί για μας, ούτως ώστε να μπορέσει μία μικρή υπηρεσία να είναι αποτελεσματική. Να σας δώσω ένα καλό παράδειγμα για την κατάρτιση. Πρόσφατα πήγαμε στην Κίνα, είχαμε την Σύνοδο Κορυφής που γίνεται κάθε δύο χρόνια ε, και ήρθαμε σε επαφές, κάναμε ένα σεμινάριο, μια ημερίδα Ε, συζητήσαμε για το πώς κατασκευάζονται οι τηλεοράσεις, ε, ε, ούτως ώστε να είναι ασφαλείς. Ασφαλείς ιδίως για τα μικρά παιδιά που τους αγοράζουν οι γονείς τους σε δική τους τηλεόραση και οι κατασκευαστές οι κατασκευαστές ενημερώνουν τους γονείς για το πώς θα βοηθήσουν τα παιδιά τους να προστατευτούν από τις επικίνδυνες επιπτώσεις της τηλεόρασης. you... Επίσης πήγαμε μαζί με τους Ευρωπαίους στην Κίνα για να μιλήσουμε για ασφάλεια. Αντί να φτιάχνουμε παγκόσμια προϊόντα, εμείς εστιάσαμε ε, στα πιο επικίνδυνα προϊόντα για τους καταναλωτές, για να έχουμε κοινές, ε, κοινά σεμινάρια, ας πούμε, σε χώρες όπως η Κίνα ή το, σεμινά, το Βιετνάμ. Τα περισσότερα παιδικά προϊόντα είναι κινέζικα, παράγονται στην Κίνα. Μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ε, τέτοιες κοινέ προσπάθειες κατάρτισης. Επίσης άρχισα να μιλάω σε κολέγια και πανεπιστήμια και να συνεργαστούν μαζί μας. Εκεί υπάρχουν καθηγητές που είναι διατεθειμένοι να πάρουν άδεια από τη δουλειά τους για να πάνε στην Κίνα ή στο Βιετνάμ. Και με αυτόν τον τρόπο συνεργάζονται μαζί μας και προωθούν την κατάρτιση αυτές τις χώρες. Νομίζω ότι καλύτερα η πρόληψη παρά η θεραπεία. Αν μπορούμε να προλάβουμε λοιπόν τους τραυματισμούς, ε, νομίζω ότι και οι κατασκευαστές θα εποφεληθούν, γιατί μακροπρόθεσμα είναι λιγότερο δαπανηρό να δραστηριοποιηθούν σε επίπεδο πρόληψης. Ειδικά α, κατασκευαστές μικροί, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ας πούμε, που δεν έχουν δικηγόρους, μεγάλο δικηγόρους, να τους εξηγήσουν, ας πούμε, όλα τα θέματα τα νομικά. Ελπίζω να σας απάντησα. Ναι. Η κυρία Στάιλερ, τελευταία χρόνο έχουμε. Έχουμε μέχρι τις 6.30 αν δεν απατώ με την αίθουσα. Αν θέλετε να κάνουμε και δεύτερο γύρο και παραπάνω, αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις. To um, raise further questions while we have the great opportunity to talk to you. Uh, so, Mrs. Styler. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Mrs. Tenenbaum, for your η κυρία Στάιλερ, ευχαριστώ κυρία Τένεμπαουμ που ήρθατε σήμερα εδώ να μας μιλήσετε. Πολύ διαφωτιστικό και ενημερωτικό ε, και... και στη Σκοτία Πραγματικά ε, κάποιος πέθανε, επειδή πέθανε ακριβώς από, ε, γιατί κρεμάστηκε στο σκηνή κατεβάζοντας τις γρίλες σε ένα παράθυρο. Πολύ σημαντικό αυτό. Και υπάρχουν και απλές λύσεις από το design ε, και από το σχεδιασμό και το έχουμε συζητήσει και στη Σκοτία πώς μπορούμε να πείσουμε τους κατασκευαστές. Δεν είναι σκοτσέζικο το θέμα, αφορά όλο τον κόσμο για να σχεδιάζονται διαφορετικά τα προϊόντα, να είναι πιο κίνδυνα. Πρόσφατα πήγαμε στο Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης. Θεωρείτε ότι τα διεθνή πρότυπα είναι ε, αποδοτικά. Καλό είναι να συζητούμε για τα πρότυπα που έχουμε ο καθένας, αλλά να δούμε και πώς χαράσουμε διεθνή πρότυπα. Εγώ είμαι ε, ε, η συγκήτρια για προϊόντα κατασκευαστικά υλικά. Ναι, γιατί θέλουμε να δούμε και την προστασία ε, όχι μόνο των καταναλωτών και των εργαζομένων στις οικοδομές. Αυτό το θέμα είναι στη δική σας αρμοδιότητα. Και μετά, Πώ κατασκευάζονται τα σπίτια, α πούμε. Τι γίνεται στην ασφάλεια, την πυρασφάλεια των σπιτιών ή την προστασία από το μονοξίδιο του αζότου ή ε, από τις πίθες, ε, από τις, ή, τους κατεοριστήρες, Η Κρίστερ Σάλντε Μόσε προηγουμένω μίλησε για τα προϊόντα, αλλά δεν είναι μόνο τα φυσικά προϊόντα, τα υλικά προϊόντα, με τι υπηρεσίε τι γίνεται. Κάποια προϊόντα υπηρεσιών, πώς παρέχονται αυτά και πώς ε, ενημερώνεται τους καταναλωτές στην Αμερική. Το συζητούμε πάρα πολύ αυτό τον καιρό εδώ και θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσουμε και τις δικές απόψεις. Και είναι πολύ αξιόλογη πραγματικά η προσπάθεια που κάνετε, η πρωτοβουλία σας και θέλω να μας ε, ενημερώσετε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Ε, τώρα, ε, το θέμα με τις χρήλες στα, στα παράθυρα. Πώς συνεργάζονται ο Καναδάς με τις Ηνωμένε Πολιτείε για να εκδώσουμε μια κοινή δήλωση. Να υπάρχει μια προδιαγραφή, ένα πρότυπο που να το υιοθετήσουμε για να προστατεύουμε τα παιδιά. Μπορούμε να το κάνουμε αναπερίπτωση αυτό, εφόσον υπάρχει προθυμία και βούληση να συνεργαστούμε. Και νομίζω ότι υπάρχει, το έχουμε δει επανειλημμένο αυτό. Αναπροϊόν, έτσι. για ένα πρότυπο ε, για ουσίες, για το μόλυβδο για το ε, κάδμιο. Ε, αλλά για τα ρολά των παραθύρων και τις γκρίλης. Ε, τώρα τα διεθνή πρότυπα. Ε, η αγορά είναι παγκόσμια. Όταν κατασκευάζει μια εταιρεία κάτι στην Κίνα, θέλει να το πουλήσει παντού, σε όλο τον κόσμο. Είναι δύσκολο δηλαδή να έχεις άλλες προδιαγραφές για τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλες για εδώ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένες πολιτείες έχουν αυστηρότερες προδιαγραφές από την ε, ε, ομοσπονδιακή νομοθεσία. Πρόσφατα αγόρασε ένα χλοκοπτικό μηχάνημα και γράφει ε, να, δεν, να μην πωλείται στην Καλιφόρνια γιατί έχει υψηλότερε προδιαγραφές. Και η Καλιφόρνια πάντα άνοιγε το δρόμο ε, σε θέματα προστασίας των καταναλωτών. Και άλλες φορές έχουν εκείνη πιο αυστηρό πρότυπο ε, από άλλες πολιτείες. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κάπου ορισμένοι επιστήμονες που θεωρούν ότι η προδιαγραφή πρέπει να είναι αυστηρότερη. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζονται και επιστήμονες λοιπόν σε αυτό το θέμα, ε, να υπάρχει διεθνής επιστημονική συνεννόηση για τους κινδύνους από τα προϊόντα. Ας πω, το κάναμε για τις φθαλικές ενώσεις στο πάνελ αυτό. Καλό είναι λοιπόν να συνεργάζονται και οι επιστήμονες και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να προχωρήσουμε και στην εναρμόνιση. Οικοδομικά υλικά. Ε, πρόσφατα το ε, κοιτάξαμε αυτό για ένα ε, θέμα ενός κινέζικου προϊόντος που δημιουργούσε διάβρωση στα καλώδια στις νότιες ε, ε, πολιτείες, στη Λουιζιάννα και τη Φλόριντα. Ήταν ένα στοιχείο που υπάρχει στον τοίχο. Ε. χαλούσαν τα κλιματιστικά, τα συστήματα πυρασφάλειας και συναγερμών και αφού το ψάξαμε πολύ και με επιστημονικά στοιχεία διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ανομαλία. Και τι ήταν αυτή. Ορισμένα προϊόντα στεγνωτικά της βαφής ε, που ήταν σε λιγότερο από 5.000 σπίτια στέγνωναν ε, πολύ πιο γρήγορα το ε, υδροθρόθιον από ό,τι τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Αμερική. Γιατί έχει να κάνει με το πόσο βάρος υγρού προϊόντος ε, ε, αντέχει και ε, σε ποια αναλογία να με το γύψο αυτό το προϊόν. Λοιπόν, θα έρθουμε σε επαφή με τους Κινέζους λοιπόν, παραγωγούς αυτής της ουσίας για να δούμε πώς μπορούν να, να το βελτιώσουμε και να μοιραστούμε λίγο ε, την ευθύνη και την οικονομική. Έχει γίνει αγωγή που κοστίζει 2,6 εκατομμύρια. Ε, εφτά είναι οι ιδιοκτήτες των σπιτιών στη Βερζίνια. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε παγκόσμια αγορά πρέπει να δούμε και την παγκόσμια ευθύνη. έτσι για να προστατεύονται και να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τα προβλήματα, τα προβλήματα αυτά. Είναι σημαντικό το θέμα και μεγάλο. Και διεθνές όντως. Πυροσφάλεια. Βεβαίως. Κοιτάμε τις γεννήτριες. Ανησυχούμε πολύ γιατί ε, η πυρκαγιά είναι μεγάλος κίνδυνος. Επίσης, ε, η δηλητηρίαση από το μονοξίδιο του θείου ε, για τα συστήματα κατά του άνθρακα για τους κατονιστήρες, ε, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και είναι θέμα διεθνών προδιαγραφών και αυτό για να έχουμε το υψηλότερο πρότυπο. Ακριβώς γιατί είναι και έφλεκτα τα υλικά 16 χρόνια το δουλεύουμε αυτό και είναι και προτεραιότητα και της παλιάς ε, διεύθυνση και τη δική μας. Οι γεννήτριες ας πούμε και ε, η δηλητρίαση από μονοξίδιο του ε, άνθρακα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα κοιτάμε. Και τα πυροτεχνήματα, τους αναπτήρες, έπιπλα σας είπα για τις γεννήτριες, το μονοξίδιο του άνθρακα, όλα αυτά τα θέματα. Good. Um, got uh, one or two questions, um, but... Και εγώ μια-δυο ερωτήσεις, uh, αλλά υπάρχει και ένας άλλος ομιλητής. Ποιος θέλει πρώτος, θέλετε εσείς πρώτος. Ήθελα να χρησιμοποιήσω το προνόμιο του Προέδρου να κάνω και εγώ τις ερωτήσεις μου, αλλά ξεκινήστε εσείς. Καταλαβαίνω ότι τα φάρμακα δεν είναι στην δικαιοδοσία σας, δεν είναι αρμοδιότητά σας. Εδώ στην Ευρώπη τα πάμε καλά με τις επιθεωρήσεις ε, των εγκαταστάσεων των φαρμακοβιομηχανιών. Γιατί ο τρόπος παραγωγής των φαρμάκων είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων. Η ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων είναι Είναι πολύ σημαντικό θέμα και ε, η ερώτηση μου είναι η εξή. Εσείς ασχολείστε με την κατάρτιση, με τη διδασκαλία, προσπαθείτε με την πυθό να εκπαιδεύσετε τον κόσμο. Πηγαίνετε όμως επί τόπου να επιθεωρήσετε τις εγκαταστάσεις ε, των βιομηχανιών. Πηγαίνετε επί τόπου. Ζητώ συγγνώμη που ενδεχομένως κάνω φελή ερωτήματα, αλλά επειδή ήρθα πολύ αργά, δεν ξέρω ακριβώ τι έχετε συζητήσει και μπορεί να σα κάνω τι ίδιες ερωτήσεις με προλαλήσαντε. Ε, σας ευχαριστώ που ήρθατε, λέει η Αμερικανίδα φιλοξενούμενη. Όχι, εμείς δεν ε, επισκεπτόμαστε εργοστάσια. Αν κάποιος κατασκευαστής στις Ηνωμένε Πολιτείε, ε, ο οποίος ξέρουμε ότι επίτηδες ε, αγνοεί τους κανόνες ή τους ε, παρακάμπτει, μπορούμε να κάνουμε μια επιτόπου επιθεώρηση, αλλά συνήθως δεν το κάνουμε. Χαίρομαι που ο κύριος Κάμπος έθεσε το θέμα γιατί έχω και μια σχετική ερώτηση. Για κάπως φιλοσοφική προσέγγιση για τα παιχνίδια και για την επιτήρηση της αγοράς και την εκτίμηση της συμμόρφωσης, θα έλεγα ας πούμε έτσι. Έχετε δίκιο που δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ότι οι υπεύθυνοι κατασκευαστές πρέπει να εποπτεύουν ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής του προϊόντος. Για παράδειγμα, και τα ε, χρώματα, οι βαφές με μολύβι, με περιεκτικότητα σε μόλυβδο που δεν είχαν ελεγχθεί. Η όλη, το όλο θέμα της αποτίμησης, της συμμόρφωσης, ότι δηλαδή οι κατασκευαστές πρέπει να αποδεικνύουν έτσι ώστε να ικανοποιήσουν τις αρχές ότι είναι σε θέση να παράγουν αγαθά κατάλληλης ποιότητας που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφέ. Αυτό μου φαίνεται εμένα πάρα πολύ σημαντικό. Η διαφορά στην νοοτροπία είναι πόσο μέρος της έρευνα, του τεστ μάλλον, γίνεται από τρίτους φορείς. Αυτό είναι ενδιαφέρον να συζητήσουμε και έχουμε συζητήσει και μαζί σας και πριν. Γιατί η οδηγία για τα παιχνίδια, όταν συζητούσαμε την οδηγία για τα παιχνίδια, είχαμε συζητήσει και αν θα κάνουμε υποχρεωτική ε, εξέταση και από τρίτους φορείς. Και η άποψη που επεκράτησε τελικά στο Κοινοβούλιο, αν και δεν ήταν άποψη όλων, είναι ότι θα πρέπει οι κατασκευαστές να έχουν εργαστήρια εξέτασης των προϊόντων που θα είναι τουλάχιστον το ίδιο ικανοποιητικής ποιότητας όπως των τρίτων φορέων. Θα ήθελα να μάθω εάν θεωρείτε ότι στο μέλλον ενδέχεται να εξτάσετε πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη πέραν τώρα της θεωρίας γιατί φαίνεται να υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διαφορά προσεγγίσεων εν προκειμένου. Πάντως, κοιτάξτε, επιτρέπουμε να κάνουν τα τεστ αυτά οι ίδιες οι αλλά το εργαστήριο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο. Η Ματέλ έχει τα δικά της εργαστήρια, όπου εξετάζουν στα εργαστήρια αυτά τα παιχνίδια που φτιάχνουν, αλλά πρέπει να είναι ξεχωριστά τα εργαστήρια αυτά από την ε, ε, πλευρά του εργαστασίου από το τομέα του εργαστασίου που κατασκευάζει τα παιχνίδια και αυτό λέμε δηλαδή να είναι ένα είδος στεγανού τείχου που δεν μπορεί να διαπεραστεί. Επίσης πρέπει να έχουν διαδικασίες που αν οποιοδήποτε θεωρήσει ότι πιέζεται για να αλλάξει τα αποτελέσματα ενός τεστ να έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στην Επιτροπή Ασφάλειας Προϊόντων Καταναλωτή και να κάνει καταγγελία. Εάν λοιπόν τώρα τα εργαστήρια αυτά είναι ξεχωριστά, είναι στεγανά και δεν υφίστανται απολύτως καμία επιρροή ή πίεση από την κατασκευαστική πλευρά οι εργαζόμενοι στο εργαστήριο αυτό και μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην CPSC εφόσον σας ασκηθεί κάποια πίεση. Εάν λοιπόν υπάρχουν αυτές οι εγγυήσεις, τότε μπορεί ο κατασκευαστής να έχει το εργαστήριό του. Αλλά μπορεί να είναι και ανεξάρτητα ιδιωτικά. Τώρα έχουμε και στην ιστοσελίδα μας μια πρόταση για το τι είναι ένα εύλογο πρόγραμμα τεστ που δεν αναφέρεται μοναχά στην πρώτη φουρνιά των προϊόντων, παιχνιδιών ή άλλων, αλλά γράφουμε και ένα πρόγραμμα έτσι ώστε ο κατασκευαστής να έχει ένα πρόγραμμα που να εξετάζει τι δουλειά, αν έχει κάνει πραγματικά καλή δουλειά το εργαστήριό τους. Και τώρα για προϊόντα που δεν απευθύνονται σε, παιχνίδια, σε παιδιά, συγγνώμη, βασίζονται σε τεστ από τρίτους φορείς. Αν για παράδειγμα κάποιος κατασκευάζει ένα παιδικό προϊόν και έχει ένα εύλογο πρόγραμμα τεστ μέσα στην ίδια του την επιχείρηση, όπου κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλίζει ο κατασκευαστής πάντα ότι λειτουργούν τα τεστ αυτά. Εάν υπάρχει αυτό, αν το έχει αυτό, ή πάλι εάν προσφέρει τις υπηρεσίες ενός τρίτου φορέα, τρίτου εργαστηρίου, υπάρχει αυτή η προφύλαξη. Εάν έχει ένα εύλογο πρόγραμμα, λοιπόν δεν χρειάζεται να κάνει το τεστ περισσότερο από κάθε δύο χρόνια. Α, με αυτόν τον τρόπο χαμηλώνουμε το κόστος του κατασκευαστή και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε και την κοινή λογική αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε ώστε οι κατασκευαστές να μην αναλαμβάνουν περιττό κόστος. Αν εσείς θελήσετε πάντως να κάνετε κάτι τέτοιο, μπορείτε να υποφεληθείτε από όλη την πρώτη εργασία που έχουμε κάνει εμεί, τι συζητήσει, την έρευνα και να εξετάσετε ε, πώ έχουμε διαρθρώσει την νομοθεσία μας αυτή. Αυτό το, αυτά τα τεστ είναι περίπλοκη υπόθεση. Και μία από τις ερωτήσεις που ξέχασα να απαντήσω προηγουμένω. Αν εξετάζουμε τι ιδιωτικέ πωλήσει, τα garage sales όπως λέμε. Οι πιο πολλές πολιτείες έχουν έναν ειδικό φορέα, έναν ειδικό οργανισμό ασφάλειας προϊόντων που εξετάζει και αυτές τις ιδιωτικές πωλήσει. Εμείς δεν θα πάμε να εξετάσουμε τον καθέναν που πουλάει στην αυλή του ή στον καράζ του ε, κάποια ε, πράγματα. Το καλύτερο βέβαια είναι να ενημερωθεί ο κόσμος. Έχουμε την ιστοσελίδα του CPSC, όπου μπορεί να δει ο κόσμος τι ε, απαιτείται. Κάνουμε και εκστρατείες μέσω των μέσων, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, για να γνωρίζουν οι άνθρωποι περί τίνος πρόκειται. Συνεργαζόμαστε και με τις πολιτείες, ώστε να κατανοήσουν. Κάναμε και μια εκστρατεία μόλις το προηγούμενο καλοκαίρι όταν άρχισε ο κόσμος να κάνει αυτές τις ε, ε, πωλήσει. Ε, και είπαμε προσέχτε, προσέχτε γιατί μπορεί να παρισφρήσει ανάμεσα στα είδη που θέλετε να πωλήσετε και κάποιο προϊόν που έχει ανακληθεί. Για παράδειγμα, οι παιδικές κούνιες, τα παιδικά, τα παιδικά κρεβατάκια τα οποία περνάνε από παιδί σε παιδί και έχουμε συστήσει τον κόσμο να μην το κάνει αυτό. Γιατί υπάρχει κίνδυνος ε, να πεθάνουν παιδιά. Ε, μικρά βρέφη μέσα σε, αυτή την, ε, σε αυτές τις Σοβαρή προειδοποίηση αυτή και για μένα που είμαι παππούς. Παλιότερα βέβαια πέρασα τις κούνιες αυτές από παιδί, από παιδί σε παιδί. Πρώτα ήμουν αγωνιό, βέβαια. Α, αυτό ε, σας συνιστούμε να μην το κάνετε. Μην κάνετε τα ίδια λάθη, δηλαδή μην τι επισκευάζετε τις κούνιε με μονοτικές ταινίε και τέτοια. Κάτι ακόμα. Γιατί κάθε και εγώ έχουμε παρόμοιες εμπειρίες για τα προϊόντα, για τα έπιπλα μάλλον. Στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουμε τους αυστηρότερους κανόνες ε, για μαλακά έπιπλα τα οποία να μην, να μην ε, κινδυνεύουν από φωτιά, από πυρκαγιά και λόγω τοξικότητας. με, τον τρόπο αυτό έχουμε επιτύχει να υπάρξει κάποια πρόοδος, να αποφευθούν θάνατοι. Η ερώτησή μου, η ευρύτερη ερώτησή μου τώρα είναι πρώτα η αναζήτηση νέων ιδεών για την ε, ε πρόθεση της παραγωγής επιβραδυντικών ουσιών για τα προϊόντα αυτά. Ίσως είναι και αυτός ένας τομέας που μπορούμε να ε, αναζητήσουμε κάποιες λύσεις κοινέ. Δεύτερον, για τα ρόλα, οι ε, κουρτίνες. Είχαμε ελπίσει να υπογράψετε σήμερα και να μπορέσετε να μας ανακοινώσετε στην παρούσα συνεδρία, αλλά ίσως γίνει αυτό μέχρι τέλος της εβδομάδας. Θα είναι όμως ένα θαυμάσιο βήμα προς τα εμπρός. Ένα από τα θέματα πάντως που ίσως εξετάσουμε μέσα στα πλαίσια της, ε, της ε, διαδικασία εναρμόνισης, εάν υπάρχει κάτι κατεπήγον δηλαδή. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες συσκευέ εντό εισαγωγικών που υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολύ καιρό. Και ειδοποιούμε με εκστατείε του γονιούς ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Και το ίδιο ισχύει και για το μίσο που μπορεί να προκύψουν κάποια νέα, κάποιες χημικές συνθέσεις κλπ. όταν συναντήθηκα με την ASTM που κάνουν μεγάλες διαβουλεύσεις και επιζητούν συνένεση και βέβαια να ζητούν μια σωστή ισορροπία. Τι σκέπτεστε λοιπόν για αυτά. Γιατί αυτά θα είναι και κάτι άλλο που θα μας απασχολήσει. Όταν προς το τέλος ε, του χρόνου θα φτάσουμε να ολοκληρώσουμε την νομοθετική μας προσπάθεια εδώ στην Ευρώπη. Αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στην Επιτροπή γιατί είναι πολύ αργή η διαδικασία αυτή. Η εναρμόνιση είναι απίστευτα αργή διαδικασία. Κανένας μας λέει όχι στην εναρμόνιση, την επιθυμούμε, αλλά χρειάζεται μεγάλες προσπάθειες. Ε, ε, κάποιος να το προωθεί αυτό το θέμα. Και κάθε μία από τις διοικήσεις. Είναι σαν να χρειάζεται μια ομάδα ανεξάρτητη να επιφορτιστεί με αυτή τη δουλειά για να προχωρήσει, για να προοδεύσει και σε αυτή η υπόθεση. Γιατί εμείς δεν έχουμε ανθρώπους που να ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό, πλήρους απασχόλησης. Και μπορούν ε, να συνεργάζονται, αλλά έχουν ε, και άλλα επιμέρους καθήκοντα, γι' αυτό καθυστερεί. Δεν ε, είναι θέμα βούλησης, η βούληση είναι δεδομένη. Το θέμα της κοινή έρευνας. Ε, πολύ σημαντικό επίσης. Αν έχετε κάνει έρευνα, μοιραστείτε παρακαλώ μαζί μας τα αποτελέσματα και εμείς αντίστοιχω για να διευκολύνουμε την κατάσταση. Έχουμε τόσους πολλούς ομοσπονδιακούς οργανισμούς στις ΗΠΑ που κάνουν τόσο περισσότερη έρευνα από εμάς το Εθνικό Ερευνητικό Ίδρυμα, Επιστημονικό Ίδρυμα, το Κέντρο για την ε, Πρόληψη και Αναφορά Νοσημάτων. Εκεί έχουν πολύ περισσότερη δυνατότητα και άλλα ερευνητικά ιδρύματα από εμάς. Για παράδειγμα, το μονοξίδιο του άνθρακα ή ε, ε, τα έφλεκτα έπιπλα ε, βεβαίως μπορούν να ενταχθούν στην ίδια ομάδα δράσης, να συλλεγούν όλα τα στοιχεία όλα τα επιστημονικά δεδομένα, να συνεργαστούν πρώτα οι επιστήμονες. Να δούμε πώς έχει βιβλιογραφία, οι κύριες μελέτες και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και ας πούμε επίσης τα λουστραρισμένα έπιπλα που είναι έφλεκτα. Έτσι κάποιες ιδέες σας δίνω. Αν υπάρχουν και άλλες. Ρίτσαρτ Ματ, ε, έχετε τίποτα να προσθέσετε. Αλλά, ξέρετε, ε, τα πάντα είναι η εφαρμογή. Εκεί είναι το ζήτημα, όχι η αντίσταση για την εναρμόνιση. Δεν είναι ότι υπάρχει βούληση. Είναι τόσα τα προϊόντα και τόση έρευνα και επιστήμη να δούμε, να συνεργαστούμε σε λίγα αρχικά ε, προγράμματα και να δούμε πώς θα προχωρήσουν. Ευχαριστώ. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ε, ως άμεση συνέπεια της σημερινής συνεδρίασης ότι μας ακούει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι παρούσα να δούμε αυτό το θέμα ε, για τα έπιπλα. Είχαμε μια συνεδρίαση με πυροσβέστες την περασμένη εβδομάδα και το θέμα των φθαλικών ενώσεων σημαντικό καλέσαμε από το Ηνωμένο Βασίλειο και εσείς καλέσατε από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία ε, στο δικό σας πάνελ για να συζητήσετε αυτά τα θέματα. Ε, έχω και άλλη ε, μια ερώτηση της κυρίας Χάιντι Ρούιλε που συμμετείχε και στην προηγούμενη επίσκεψη και ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ. Ήταν και η συγκήτριά μας για τα θέματα αυτά. Χάιντι, παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση και εγώ θα πω στα γερμανικά όμως. Ich mich auch noch mal Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι. Δυστυχώς καθυστέρησα. Καθυστέρησα, λέω, γιατί ε, έχουμε προβλήματα πτήσεων αυτό το καιρό και ε, δεν μπορούμε να φτάσουμε στις Βρυξέλλες. Έχω μια συμπληρωματική ερώτηση τώρα. Κάτι που μας απασχολεί τώρα όλους είναι το θέμα ε, της τυποποίησης και των προδιαγραφών. Και ακριβώς επειδή είναι βραδία η διαδικασία, μας απασχολεί πώς θα μπορούσε να επιταχυνθεί. Σωστά κατάλαβα αυτό που λέτε, ότι και για τις ε, προδιαγραφές, απευθύνεται στους αρμόδιους οργανισμούς και ζητάτε για συγκεκριμένα σημεία να σας παρουσιάσουν προτάσει. Δεν το έχω καταλάβει. Θα με ενδιαφέρε γιατί για μας πραγματικά είναι πάρα πολύ αργή αυτή η διαδικασία και δεν έχουμε και αρκετές προφορίες για τα ενδιάμεσα στάδια. Υπάρχει και έλλειμμα διαφάνειας εκεί. Το ξέρω ότι είναι εθελοντική διαδικασία ε, και καλό είναι, ούτε θέλουμε να αποτρέψουμε κανένα, αλλά και ούτε κανείς επιθυμεί ε, καθυστερήσεις, αλλά πώς μπορούμε περισσότερο να επηρεάσουμε και τα πράγματα. Um, uh, Ο Ρίτσαρντ Ομπράιεν μου έλεγε ότι οι συζητήσεις του προσωπικού ε, είναι πολύ συχνές και έντονες. Συζητούν λοιπόν για το πώς μπορούν να τυποποιήσουν κάποια πράγματα ε, και γίνεται τώρα πολύ πιο συχνά αυτό από ό,τι στο παρελθόν. Πριν από χρόνια δεν προσπαθούσαμε να εναρμονίσουμε. Ο καθένας, ε, κάθε χώρα για το δικό της πρότυπο. Τώρα, λόγω της παγκοσμιοποίησης αγοράς, είναι σημαντικό να ανταλλάσσουμε και πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές και την έρευνα που κάνουν οι επιστήμονες, ούτως ώστε να πετύχουμε το υψηλότερο δυνατό πρότυπο ε, σε όλες τις χώρες και σε όλες τις περιφέρειες, σε όλες τις περιοχές του πλανήτη. Επίσης, έχετε δίκιο που λέτε ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ χρονοβόρα. Τα συζητάμε από σεμινάριο σε σεμινάριο, αλλά το θέμα είναι ότι μπορούμε να εστιάσουμε, να παίρνουμε ας πούμε τα ρολά και τα, τις γρίλες ας πούμε και προσπαθούμε να αρμονίσουμε ε, τα πρότυπα σε αυτόν τον τομέα. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύουμε τις Διεθνείς Επιτροπής με την ε, Επιτροπή Διεθνών Προτύπων. Προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό πρότυπο στα εθελοντικά, σε εθελοντικό επίπεδο. συζητούμε μαζί, ακούνε τα αιτήματά μας ε, για να φτάσουμε στο υψηλότερο δυνατό πρότυπο. Συμφωνώ ότι αυτές οι συζητήσεις είναι πολύ επικοδομητικές ε, και πολύ σημαντική προσπάθεια για την εναρμόνιση των προτύπων. Πριν κλείσουμε τη συνεδρίαση, βλέπω ότι έχουμε και την εκπροσώπηση εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει μια παρέμβαση και Επιτροπή, όχι κατά ανάγκη να δώσει απαντήσεις, αλλά να μας πει και αυτή την άποψή της. Ε, δεν θέλω να σας τέρισω την ευκαιρία να μιλήσετε κι εσείς. Να... Ευχαριστώ. Ε, είμαι ευγνώμων προς την κυρία Τένεμπο και τους συναδέλφους από την Επιτροπή την Αμερικάνικη Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων. Πριν από τρία-τέσσερα χρόνια Ε, μιλούσαμε για τα κοινά μας ε, προβλήματα. Τώρα ανταλλάσσουμε πέρα από τα προβλήματά μας και πληροφορίες. Πήγαμε μαζί στην Κίνα, ε, οργανώσαμε αυτά τα σεμινάρια από κοινού στην Κίνα. Νομίζω ότι είναι καλά παραδείγματα συνεργασίας. Επίσης για νέα θέματα, νέα προβλήματα που ανακύπτουν, όπως ας πούμε για τις γρίλες, συνεργαζόμαστε είπε με μία ευρωβουλευτής ότι είναι πολύ σημαντική η διεθνή συνεργασία και πολύ φιλόδοξη. Ναι, κάναμε πολλές προσπάθειες και ελπίζω ότι οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ανταλλαγή πληροφοριών που ξεκίνησε θα μας οδηγήσει στην επόμενη φάση. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όλες αυτές οι προσπάθειες που ξεκίνησαν πριν από λίγα χρόνια έχουν δώσει πραγματικά καρπούς. Και περιμένω ακόμα περισσότερους. Δεύτερο σχόλιο. Από αυτά που ακούσαμε σήμερα, όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα για μας, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την αναθεώρηση της οδηγίας ασφάλειας των κανονικών προϊόντων. Ε, χαιρόμαστε που η Επιτροπή σας, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτά τα θέματα ε, και ενδιαφέρεται για την αποτελεσματικότητα των κανόνων. Ε, η τυποποίηση των προτύπων είναι μια χρονοβόρα διαδικασία στην Ευρώπη. Ε, και χρονοβόρα διαδικασία και δύσκολη είναι η εποπτεία της αγοράς. Όταν ε, κάνω παρουσιάσεις σε διάφορα κράτη-μέλη, που το κάνω και εγώ και οι συνάδελφοί μου τακτικά, ε, ακριβώς αυτό έχω στο μυαλό μου. Ε, το 1997 είχαμε τρεις προτεραιότητες. Εφαρμογή της νομοθεσίας, εφαρμογή της νομοθεσίας, εφαρμογή της νομοθεσίας. Με αυτό το πνεύμα πηγαίνω, ας πούμε, στις προσ... σε αυτά τα σεμινάρια που κάνω και στις ομιλίες που δίνω. Όλα αυτά λοιπόν θα τα έχω υπόψη μου. Θα έρθω και σε επαφή με την κυρία Σαλντεμόζα για την αναθεώρηση τη οδηγία για την ασφάλεια των κανονικών προϊόντων. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. σε λίγες εβδομάδες θα υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία για την ανταλλαγή πληροφοριών με τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ αποφελέ για τι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Ηνωμένε Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ανταλλάσσουν πληροφορίε για την έρευνα των προϊόντων. Πληροφορίε και έρευνα. Θα έχουμε κοινή, κοινή εφαρμογή λοιπόν. μάλλον είναι ένα λιθαράκι στην πορεία για την κοινή εφαρμογή, για την αρμόνιση και τα κοινά πρότυπα. Επίσης, τον Οκτώβριο θα είμαστε μαζί στην Κίνα ε, σε μια τριμερή συνάντηση στη Σανγκάη, στην έκθεση της Σανγκάης. Ευρώπη, Ηνωμένε Πολιτείε, Κίνα. Σε αυτή την τριμερή συνάντηση. Και θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις για επαφές με Κινέζους και άλλους ε, για να προωθήσουμε την μας, το κοινό μας στόχο που είναι η ασφάλεια. Σας ευχαριστώ που είχα εγώ και τα μέλη της Επιτροπής να έρθουμε εδώ με τον πρόεδρο, σε αυτή την Επιτροπή μαζί με τον πρόεδρο Χάρμπορ για να προωθήσουμε τα θέματα ασφάλειας και ελπίζω τα επόμενα χρόνια να συνεργαστούμε ούτως ώστε να προωθήσουμε από κοινού την ε, ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων προς το καλό των ε, Αμερικανών και Ευρωπαίων καταναλωτών. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Ευχαριστώ. Και εγώ, κυρία Πρόεδρε, εξ ονόματος ε, της Επιτροπής μας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Τέρμπαου και ε, σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να έρθετε να μας μιλήσετε. Περίπου δύο ώρες, πολύ χρήσιμη και πολύτιμη ανταλλαγή απόψεων και πέρα από διάφορε πολιτικές ομάδες ε, όλοι οι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο ενδιαφέρονται πάρα πολύ και είναι πολύ προσιλωμένοι στο έργο αυτό της προστασίας των καταναλωτών και βεβαίω ενδιαφερόμαστε πολύ ε, η ασθενή συνεργασία με άλλους νομοθέτες, Κοινοβούλια των Κρατών Μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω εκτελεστική εξουσία και θα σας ενδιαφέρει να μάθετε πιστεύω πώς ε, είναι η προσήλωση των εκλεγμένων ε, εκπροσώπων των Ευρωπαίων. Αλλά και οι ε, ψηφοφόροι μας απευθύνονται σε εμά όταν έχουν τέτοια ζητήματα και είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας και τη διεθνή διάσταση αυτής της συνεργασίας. Και τέλος, χαίρομαι που ήταν παρόν ο συνάδελφος κύριος Μορέρ εδώ, γιατί ε, να έχουμε καλές και βελτιωμένες προδιαγραφές προστασίας καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο εξαρτάται και από τη συνεργασία μας με τις ΗΠΑ και την εθάρρυνση του παγκοσμίου και του διεθνούς εμπορίου με όσο γίνεται υψηλές προδιαγραφές. Και θα ήθελα να ξαναπώ αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι η αγορά ε, είναι παγκόσμια και θέλουμε να έχουμε παγκόσμια αγορά με ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε ήδη και στην Ευρώπη και στι ΗΠΑ. Και όσο περισσότερο συνεργαζόμαστε, τόσο ε, μεγαλύτερο θα είναι το όφελος για τους συμμετέχοντες και τους κατασκευαστές που στο κάτω-κάτω δημιουργούν και θέσει απασχόληση σε όλο τον κόσμο αλλά και για τους καταναλωτές που αγοράζουν τα προϊόντα αυτά. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά μας ε, να σας υποδεχτούμε σήμερα εδώ. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι και προσκεκλημένοι ε, να ξανάρθετε σε επόμενη επίσκεψή σας στην Ευρώπη. Πολύ χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην μελλοντική σας ε, εργασία. Θα σας δω και την Παρασκευή στη διάσκεψη της Ισπανικής Προεδρίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα διοργανώσει τέλη Οκτωβρίου, είπατε, ένα σεμινάριο στη Σανγκάη. Ε, και βλέπουμε λοιπόν και την παγκόσμια διάσταση εκεί. Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να εκπροσωπήσω το κοινοβούλιο και εκεί. Με κανένα δυο συναδέλφους ενδεχομένως. Και αυτό θα είναι καλή ευκαιρία να τα ξαναπούμε για να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και με την Κίνα. Το Μάρτιο του 2008 η Επιτροπή μας πήγε στη Σανγκάη και έχουμε αντίστοιχη προσέγγιση με τη δική σας και παίρνουμε πολύ σοβαρά τις ευθύνες μας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και πάλι και θέλω να πω επίσημα στα μέλη της ε, Επιτροπή μας σε η επόμενη συνεδρίαση θα είναι στι 23 και 24 Ιουνίου. Στι 23 τι ώρα είναι μια στιγμή στις... Το πρωί είναι. Το πρωί έχουμε για τα... μια ακρόαση για την εναρμόνιση των προτύπων, για την τυποποίηση και μετά... Εν πάση 23 και 24 Ιουνίου συνεδριάζει η Επιτροπή μας